Thank Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη για τις ερωτήσεις και την υποψηφία επίτροπο για τις απαντήσεις. Πραγματικά ήταν ένα ε, δύσκολο απαιτητικό πρωινό, αλλά επίσης πολύ χρήσιμο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Πριν δώσω το λόγο στην υποψηφία επίτροπο για τις ε, καταληκτικές της ε, δηλώσεις, θα ήθελα να καλέσω τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών να κάνει μία δήλωση τριών λεπτών έτσι όπως ε, το συνηθίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της, ε, Επιτρο... Περιφερειακής Επιτροπής και κυρία Επίτροπε, Βεβαίως για μας η πολιτική συνοχή είναι πρωτεύουσα σημασίας γιατί ξέρετε ότι οι τοπικές αρχές τις οποίες εκπροσωπούμε είναι τελικά οι αποδέκτες του ε, περίπου 70% των διαφορετικών ταμείων. Η Επιτροπή Περιφερειών καλείται να διαδραματίσει το ρόλο ενός ενδιάμεσου μεταξύ ευρωπαϊκών και τοπικών αρχών. Και θα ήθελα εν συντομία να επιμείνω σε ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικά για μας. Η έκτη έκθεση για την ε, κοινωνική και εδαφική συνοχή προβλέπει ένα νέο εδαφικό όραμα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής Ευρώπη 2020 ε, και θα υπάρξει η λευκή βίβλος η οποία θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε προόδους όσον αφορά την πολιτική συνοχής και μετά το 2020. Αναφέρθηκε εδώ το πρόβλημα των αστικών περιοχών και ελέγχθη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια λευκή βίβλος, μια ολοκληρωμένη αστική ατζέντα ε, η οποία να επιτρέψει την ε, ολοκλήρωση της πολιτικής. Τα διαρθωτικά ταμεία, 350 ε, δις, θα συνεχίσουν ε, να διατίθενται. Ε, τι θα προτείνατε εσείς εκ μέρους της Επιτροπής ούτως ώστε να υποστηρίξετε μια μεγαλύτερη απορροφητικότητα των ε, πόρων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Γιατί μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα αυτό μόνον εφόσον συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ΣΑΣΑ ε, η Επιτροπή Περιφερειών ε, ζήτησε ε, να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειών και προβλέπει βεβαίως το σύμφωνο σταθερότητας στην ενίσχυση της απασχόλησης στις πιο μειονεκτούσες περιοχές. Εμείς ε, πρόκειται να ορίσουμε και να ελοπίσουμε μαζί με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την, ε, μια στρατηγική αποκεντρωμένη επικοινωνία τη Ευρωπαϊκή Πολιτική, ούτω ώστε να εξηγήσουμε στου Ευρωπαίους πολίτε την προσθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανοιχτές ε, ημέρες, οι οποίες διοργανώνουμε με την ε, Περιφερειακή Επιτροπή, συνιστούν μια μοναδική ευκαιρία για να γίνει κάτι τέτοιο. Για τις ε, γειτονικές, για χώρες ε, γιατί υπάρχουν σχέσεις με τη Νότια Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη. Εδώ η πολιτική αποκέντρωση οδηγήσε στην ενίσχυση των δεσμών με τις ε, τοπικές αρχές υπέρ της αύξησης και της δημιουργίας των θέσεων απασχόλησης. Κυρία Υποψηφία Επίτροπε, ε, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που εξαγγείλατε την ε, δέσμευσή σας να γίνετε μια πρέσβυρα υπέρ της, ε, των αστικών περιοχών και των περιφερειών. για την Επιτροπή Περιφερειών, εκ μέρους Επιτροπής Περιφερειών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που προτίθεστε να εφαρμόσετε μια αρχή την οποία και εμείς στηρίζουμε την αρχή της ε, διακυβέρνησης. Παρακαλώ. Η κυρία Κρέτσου, υποψήφια επίτροπος. Ας προβεί στην σύντομη καταλεκτική της ε, δήλωση που να μην υπερβεί τα πέντε λεπτά. Θα είμαι και συντομότερη των πέντε λεπτών, κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι μακρηγόρησα τις απαντήσεις μου. Μιλήσαμε τρεις ώρες τώρα σε τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πολιτική συνοχή. Έχω κάποιες σκέψεις ωστόσο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ήταν συναισθηματικά φορτισμένη η περίοδος αυτή των ε, τριών ωρών, αλλά ήμουν και οκτώ χρόνια εδώ. Άρχισα ένα χρόνο πριν να ενταχθεί η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρήτρια. Και θυμούμε, σαν ήταν χθε, την πρώτη μέρα που εισήλθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα συναισθήματα που με διακατήχαν όταν έγινα για πρώτη φορά ευρω, ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να σας πω ότι θα ήταν πολύ δυσκολότερο για μένα να είμαι σήμερα ενώπιόν σας χωρίς την τεράστια εμπειρία που απέκτησα στη διάρκεια των 8 αυτών ετών ως Ευρωβουλευτής. Ορισμένοι εξημών με γνωρίζετε. Όπως ήμουν θα παραμείνω. Θα ήθελα να διατηρήσω και τις ίδιες σχέσεις μαζί σας που είχαμε πάντοτε. Γνωρίζω σε ό,τι αφορά την δική σας επιτροπή τις θετικές εμπειρίες που είχαμε. Πάντοτε θα θέλω να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας και να λαμβάνουμε από κοινού αποφάσεις. Γιατί πρόκειται για πολύ σημαντικό τομέα και είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε μαζί προς το συμφέρον των πολιτών και της Ευρώπης γενικότερα. Σας βεβαιώνω ότι εάν τελικώς διοριστώ επίτροπος θα αγωνιστώ υπέρ των ίδιων αξιών υπέρ των οποίων εργαστήκαμε και μαζί ως Ευρωβουλευτές όλα αυτά τα χρόνια. Αξιοπρέπεια, ίση μεταχείριση για όλες τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και πάλι και πάντοτε θα προσέρχομαι ενώπιον σας με ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά δηλαδή που θα θέλετε ε, να με δείτε και βεβαίω όταν θα έχετε κρίνει πρώτα περί της μοίρας μου. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος Μιχαήλοβα, ευχαριστώ και εσάς κυρία Κρέτσου και όλα τα μέλη. Η συνάντηση για την αξιολόγηση των συντονιστών που θα γίνει σήμερα το απόγευμα και κλεισμένων των θυρών από τη μία μέχρι τις δύο απογευματινές ώρες στο 4Β001, αίθουσα 4Β001 και τώρα εδώ λίγη συνεδρίαση.